invitaros. Venga, pido un poquito de orden y que la gente... Ας ξεκινήσουμε παρακαλώ η ισχύα για να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Είμαστε στο σημείο 11 τη ημέρησιας διάταξης. Τροπήση του κανονισμού 302 2009 για τη θέσπιση πολιετού σχεδίου αποκατάσταση του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο. Εισηγητή κ. Ραούλ Ρωμέβα ή Ρουέδα. Δίνω το λόγο στον κύριο Ρωμέβα. Εν συντομία, να σας παρουσιάσω μία μου σκέψη. Η έκθεση αυτή έχει ως ε, στόχο να καθορίσει τη θέση του Κοινοβουλίου σε ένα θέμα το οποίο φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι είναι θέμα μεταγραφής. Το πιο απλό θα ήταν λοιπόν να υιοθετήσουμε την πρόταση της Κομισιόν, όπως υποβλήθηκε στην ICAT. Ε, όμως σκεφτήκαμε μαζί με άλλους συναδέλφους να υποφεληθούμε της ευκαιρίας για να καθορίσουμε και τη δική μας στάση ως κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό αυτό γιατί πρέπει να στείλουμε στο Συμβούλιο ένα μήνυμα. Το μήνυμα ότι είμαστε ένα αυτόνομο όργανο και διατηρεί τη δική του θέση. Είναι καλή ευκαιρία λοιπόν να γίνει αυτή η δουλειά. ακόμα και τις τροπολογίες με αυτόν τον τρόπο πρέπει να τις δούμε. Δηλαδή το κοινοβούλιο πρέπει να έχει μια αυτόνομη θέση, μια αυτόνομη στάση, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να είμαστε επικοδομητικοί. Οι τροπολογίες είναι ελάχιστες, αυτές προτείνουμε. Ε, και για ορισμένες από τις ε, τροπολογίες που υποβλήθηκαν χρειάζεται να ζητήσω αρνητική ψήφο γιατί ήταν ταυτόσιμες με τη θέση και τις προτάσεις του Συμβουλίου. Ωραία, περνάμε στις ψηφοφορίες. Η κυρία Ρόντος δεν έχει κάρτα ψηφοφορίας, υπάρχει και κανείς άλλος. Όλοι έχετε. Κυρία Ρόντος, μου λέτε τι θέλετε να ψηφίσετε. Ψηφίζουμε την τροπολογία υπαριθμών 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Του εισηγητή η τροπολογία αυτή. Λίγη ψηφοφορία. Επτά υπέρ, έντεκα κατά, ε, απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών έξι της Επιτροπής ΕΜΒΗ. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 8 υπέρ 10 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 του κυρίου Τσουκαλά. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Τι ψηφίσατε, υπέρ, υπέρ, κατά. Ο, οκτώ ψηφί υπέρ, δέκα κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 4 του κ. Κάντεκ. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 6 έχει αποσυρθεί. Περνάμε στην τροπολογία 7 της Επιτροπής ΕΜΒΗ. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 2 του εισηγητή. Άρχεται η ψηφοφορία. Se cierra la votación. Λίγη Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία υπαριθμών 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Είναι τροπολογία της Επιτροπής ΕΝΔΙ. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 του εισηγητή. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 9 της Επιτροπής ΕΜΒΗ. Έναρξη ψηφοφορίας. Λήξη. Τι ψηφίσατε κυρία Ρόντουστ. Υπέρ. Ε, ισοψηφία. Άρα απορρίπτεται και αυτή. Τροπολογία παριθμών 11 της Επιτροπής ΕΜΒΗ. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται Συγγνώμη. Ναι, μου έκανε εντύπωση. Ε, τροπολογία υπαριθμών 11. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 12 της ΕΜΒΗ. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 της Επιτροπής ΕΜΒΗ. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 της ΕΜΒΗ. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 της ΕΜΒΗ. Ψηφίζουμε. Λίγη ψηφοφορία. Τι ψηφίσατε κυρία Ρόντος, είπε. Απορρίπτεται η 10-10 ισοψηφία. Τροπολογία επαριθμών 4 της ΕΜΒΗ. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 5 της ΕΜΒΗ. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Α, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την, την νομοθετική πρόταση όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 18 ψήφοι υπέρ, μία κατά. Εγκρίνεται, υιοθετείται. Ψηφίζουμε τώρα το ψήφισμα, το νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία, ομόφωνα υπέρ. Συγχαρητήρια παρόλο που ξέρω ότι ο εισηγητής δεν είναι πολύ ικανοποιημένο. Πρέπει να ζητήσω από την, να ρωτήσω την ε, Κομισιόν να τη ρωτήσω αν δίνει τη συγκατάθεσή της ο εισηγητής να, αν δίνει την άδειά της ο, της ο εισηγητής να διαπραγματευτεί με το Συμβούλιο ε, την έγκριση πρώτη ανάγνωση του κειμένου. Ε, αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθούμε στη, σε, σε τέτοιου είδους νομοθετικά ψηφίσματα. Η Κομισιόν. Όχι, κυρία Ρέρο. Ε, στις τρεις πρώτες ψηφοφορίε είχα τεχνικό πρόβλημα και δεν μπόρεσα να συμμετάσχω. Ε, θα σα ενημερώσω γραπτός για την ψήφο μου. Δεν λειτουργήσε η κάρτα μου στις τρεις πρώτες ψηφοφορίε. Δεν αλλοιώνει το αποτέλεσμα, εντάξει. Αλλά θα ήθελα να καταγραφεί η άποψή μου. Δεν ακούμε τι λέει η πρόεδρο, δυστυχώ εκτός μικροφώνου. creo que tengo que encender. Con esto pasamos al voto siguiente. Ωραία, περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Σημείο 12. Έκθεση Φερέιρα. Μισό λεπτάκι, άσε με να μιλήσω, ας πω τι θα ψηφίσουμε και μετά θα, και μετά θα προτείνω ψηφοφορία σε μπλοκ. Δεν με αφήνετε να μιλήσω και παρόλο που εγώ μιλάω γρήγορα τροποποίηση του κανονισμού 1198-2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλία. Εισηγητή ο κ. Φερέιρα. Ο κ. Φερέιρα θέλει το λόγο. Κύριε Φερέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, δεν έχω αναφέρει στον κατάλληλο ψηφοφορία ποια είναι η άποψή μου για τι τροπολογίε. Ε, θα ήθελα να σα πω ποια είναι η άποψή μου λοιπόν για τι διάφορε τροπολογίε. Ε, συναντήθηκα με τους και ηγητές, ε, οι ίδιοι λοιπόν γνωρίζουν τη θέση μου. Θα ήθελα να σας ενημερώσω και εσάς. Δεδομένης της φύσης και του περιεχομένου της νομοθετικής πρότασης της Κομισιόν ε, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό. Υπ' αυτό το πνεύμα εργαστήκαμε Τουλάχιστον εργάστηκα εγώ στη σύνταξη της νομοδότησης. Τούτου λεχθέντος ε, θεωρώ ότι οι τροπολογίες που υποβλήθηκαν πριν από μερικές εβδομάδες από το Συμβούλιο και που προτάθηκαν ως τροπολογίες στην έκθεση ε, θεωρώ ότι ε, είναι περιτές και ακατάλληλες. Δεν προσθέτουν τίποτα. Το αντίθετο θα αποτελέσουν περιττό διοικητικό άχθος. Οι τροπολογίες αυτές ε, αντικατοπτρίζουν τη γνώμη ορισμένων χωρών του Συμβουλίου. Μια ομάδα χωρών που και στο παρελθόν ε, έχουν προσπαθήσει να αγνοήσουν τις δυσκολίες, δημοσιονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με αυτόν τον τρόπο δεν θέλουν να συνεισφέρουν στην λύση των προβλημάτων τους. Ε, δεν θα ήθελα να προτείνω κάποια για αντίθεση με αυτές του Συμβουλίου, αλλά ε, γιατί θέλω να ολοκληρωθεί η διαδικασία το συντομότερο δυνατό. Συνεπώς δεν θα διαφωνήσω με τις τροπολογίες του κ. Καντέκ. Μπορούν όλες αυτές οι τροπολογίες να ψηφιστούν ε, on block ε, ως δέσμοι. Ε, εγώ αυτό που θα ζητήσω, η δική μου θέση είναι η αποχή. Ε, ε, δυστυχώς ε, αντικατοπτρίζουν θέσεις ορισμένων χωρών του Συμβουλίου που δεν, θέσεις που δεν δέχομαι αλλά δεν θέλω να μπλοκάρω και τη διαδικασία. Ε, αυτές οι χώρες του Συμβουλίου ε, είναι αυτές που πιο πολύ θα, χρήσι, θα ωφεληθούν από τη μη χρήση, ε, την αδυναμία χρήσης των δυνατοτήτων που δίδονται ε, στις πιο αδύναμες χώρες από το, τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την μείωση της, ε, του ποσοστού συγχρηματοδότησης. Ε, χώρες, ε, πόροι οι οποίοι δεν θα χρησιμοποιηθούν από αυτές τις ε, χώρες προφανώς θα χρησιμοποιηθούν από τις άλλες χώρες που είναι αυτές οι οποίες υποβάλλουν και αυτές τις τροπολογίες. θα είναι αυτές οι ίδιες χώρες, αυτές πιο πολύ θα ωφεληθούν από τις προτάσεις αυτές. Αυτό μας εξηγεί και τα συνεχή προσκόμματα τα οποία θέτουν αυτές οι χώρες εδώ και κάποιο καιρό. Πρόεδρος. Αν δεν διαφωνεί κανένας, θα υποβάλω όλες τις τροπολογίες unblock. Τροπολογίες του κ. Καντέκ. Δεν διαφωνεί κανένας, έτσι. Άρχεται η ψηφοφορία για όλες τις τροπολογίες μαζί. Συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν ακούμε τον κύριο Ρωμέβα. Θέλετε για πολλέ ε, τροπολογίε να ζητήσετε χωριστή ψήφο. Για τέσσερι. Ποιε είναι αυτέ οι τέσσερι, Οι 15, οι, 16, οι 22, συγγνώμη, οι 6 και οι 8. Εσεί κύριε Γκάλαγκερ. Δεν θα σας δημιουργήσω πρόβλημα οι εκπρόσωποι της Άλντε θα απόσχουν για λόγους αρχής. Δεν πρόκειται να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες, το έχουμε συζητήσει ήδη παλιότερα. Ωραία. Τροπολογία 14. Τίθεται σε ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία, τροπολογίες 16 21. Άρχεται η ψηφοφορία. 16 21. Κλείνει η ψηφοφορία. Τροπολογία 22. Ψηφίζουμε. Κλείνει η ψηφοφορία εγκρίνεται. Τροπολογίες 23 ως 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 9 ως 13. Λίγη ψηφοφορία εγκρίνονται. Ψηφίζουμε την νομοθετική πρόταση όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 16 ψήφοι. Υπέρ τρεις αποχές. Ψηφίζουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη εγκρίνεται 19 ψήφοι υπέρ ομόφωνα. Συγχαρητήρια. Θα πω το ίδιο που είπα και πριν. Θα ζητήσω από την Κομισιόν να συγκατεθεί με αυτό το αποτέλεσμα ο εισηγητής να διαπραγματευτεί τη δυνατότητα ε, ολοκλήρωσης του, των διαπραγματεύσεων σε πρώτη ανάγνωση με το Συμβούλιο. Ωραία, συμφωνεί η Κομισιόν. Ο εισηγητής μπορεί να διερευνήσει την πρώτη ανάγνωση. Περνάμε στο επόμενο σημείο. 14 της ημερησίας διάταξης. Οι συντονιστέ σήμερα το πρωί αποφάσισαν να μην θέσουμε σε ψηφοφορία την έκθεση Ριβελίνη, γιατί το Συμβούλιο Υπουργών την περασμένη εβδομάδα στι Βρυξέλλε, την περασμένη Παρασκευή συγκεκριμένα, υιοθέτησε αυτή την πρόταση. Συνεπώς, έχουμε συγκεκριμένη νομοθετική πράξη και μπορούμε να ε, προσφύγουμε στο δικαστήριο. Οι συντονιστές ε, αποφάσισαν να προσφύγουμε εναντίον του Συμβουλίου στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους λαθασμένης ε, επιλογής νομικής βάσης. Ελπίζουμε ότι το Δικαστήριο θα μας δικαιώσει. Φαίνεται να έχουμε δίκιο. Έτσι μας φαίνεται μας. Ωραία. <coughs> Τι συμβαίνει. Περνάμε στο σημείο 14. No, eso eso no se puede, si no se puede votar, si vamos al Tribunal de Justicia no se puede. Bueno, que no, que no, que nada. Venga, pasamos al punto Pero no 14. Περνάμε στο σημείο 14 de ataxis. Μια Ευρώπη χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους. Η συγγήτρια κυρία Τρότμαν των Σοσιαλιστών. σχέδιο γνωμοδότησης της ηγέτριας. Παρακαλώ πολύ όσοι φεύγουν να μην κάνουν τουλάχιστον θόρυβο, γιατί οι υπόλοιποι θέλουμε να δουλέψουμε. Κυρία Συγγήτρια, έχετε το λόγο. Σας παρακαλώ. Κύριε Ρωμέβα. Κύριε Λεβίν. Ε, σαν να είμαστε σχολείο είναι εδώ. Σας παρακαλώ πολύ, ησυχία. Κυρία Τροτμάν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα θα παρουσιάσω το περιεχόμενο αυτής της εκθέσεως. Είναι μια γνωμοδότηση σε μια Ευρώπη που θα είναι αποτελεσματική στη χρήση των πόρων και τρεις παρατηρήσεις έχω να κάνω σε σχέση με τις παραγράφους οποίες έχω προτείνει. Κάνω μια ανακεφαλαίωση και θα ήθελα να το λάβετε υπόψη αυτά στο φάκελό σας. Η γνωμοδότηση που παρουσιάζεται εδώ συμπληρώνει την έκθεση του κ. Σαφάντη, ο οποίος λέει πολύ σαφώς ότι η ελεγγύη αποτελεί μέρος της στρατηγικής όσον αφορά τη χρήση των πόρων. Δεύτερη παρατήρηση, τα περισσότερα σημεία της γνωμοδότησής είναι, ήταν μέσα στα θέματα της όλης συζήτηση που είχαμε ζητήσει για την θεώρηση της κοινή πολιτικής της αλληλείας. Η πολιτική λοιπόν αυτή είναι σύντομη, είναι πάρα πολύ ειλικρινή και τι θα πρέπει η Επιτροπή αυτή της Αλληλείας να κάνει όσον αφορά την παραχώρηση, τη δυνατότητα παραχώρηση ποσοστώσεων της Αλληλείας ή του Ταμείου Αλληλείας. Τρίτη παρατήρηση, θα πρέπει να αναπτυχθεί μια καινούρια οδός όσον αφορά την κατανάλωση, τη βιώσιμη κατανάλωση, της κατανάλωσης, συγγνώμη, έτσι όπως φαίνεται στην έκθεση του προλαλήσαντος εισηγητού πράγμα το οποίο μας κάνει να περιορίσουμε την αλίευση για να συνάδει με τον οικονομικό παράγοντο, με τους παράγοντες, τους κοινωνικούς, τους περιπαντολογικούς, αλλά και μια όλο και περισσότερο αυξανόμενη κατανάλωση των αλλιευτικών προϊόντων πράγμα το οποίο δημιουργεί βεβαίω εισαγωγή όλο και περισσότερο ε, ηχθείων, αλλά και μείωση των αποθεμάτων των στόξ. Η δύο κυρία Πρόεδρε τι γενικότερε παρατηρήσει που ήθελα να κάνω σε σχέση με αυτή τη γνωμοδότηση, υπενθυμίζοντα ακόμα ότι όντω σταδιακά και βαθμιδών ε, για το RMD, στο 2, παράγραφο 2, στην παράγραφο 3, παράγραφο 4, πράγματα 6 επίσης όσον αφορά τα καύσιμα για τις μηχανές. Πολύ σύντομα δίνουν τους προσανατολισμούς, μερικούς ε, προσανατολισμούς και έρχονται να συμπληρώσουν την έκθεση του κ. Ζευκόφσκη. Ευελπιστώντας πως συνάδελφοι θα εκτιμήσουν τις προτάσεις που οποίες εγώ σας υποβάλλω. Ευχαριστώ πολύ. Sí, eh, de la, por parte de la comisión me han dicho que está, a ver... Eh. Εκ eh, Comisión της Κομισιόν είναι εδώ ο κύριος ή η κυρία Τζόνστον. Ποιος είναι? Ναι, εδώ είναι. Ο Τζόνστον. Έχετε το λόγο. Ζητώ συγγνώμη που δεν ήξερα αν ειστε αντρα άντρα ή Πολύ ένα-δύο σημεία τα πιθανά. Έχω εμπειρογνώμενε μαζί μου σε σχέση δώσαν αυτό το οδικό χάρτη που είχαν υιοθετηθεί το Σεπτέμβριο και είναι μια διαφορετική ανακοίνωση από αυτή που υιοθετήθηκε τον Γενάρη, στην οποία βασίστηκε η σημερινή γνωμοδότηση που είχαν ο μα. Αλλά επίση θα ήθελα να προσεπιστεί στο προσοχή στο γεγονό. Από τότε λοιπόν αυτή που έγινε το Γενάρη, τώρα υπάρχει μια ανακοίνωση η οποία είναι πλαίσιο ήταν αυτή τότε και τώρα υπάρχουν περισσότερε λεπτομέρειε οι οποίε έχουν εισάρθει για τη στρατηγική του 2020 όσον αφορά τη βιωσιμότητα, πράγματα που έχουν δημιουργηθεί συγγνώμη, το Σεπτέμβριο επί του θέματος αυτού. Έτσι λοιπόν υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία έχουν εισαχθεί από τότε από το Γενάρη. Θα πρότεινα λοιπόν, εάν δείτε πραγματικά το κείμενο το οποίο έχει αυτή τη στιγμή που έχει ε, εισαχθεί, βασίζεται πολύ περισσότερο στον οδικό χάρτη, ενώ από τότε υπήρξαν πολλά πράγματα τα οποία έχουν γίνει και θα πρέπει βεβαίως να λαφθά, να αντικατοπτρίζει και όλα αυτά που έχουν συμβεί από τότε. Αλλά αφήνω εδώ τους ε, παρευρισκόμενους εμπειρογνώμονες να πάρουν και αυτοί το λόγο και αν θέλουν να προσθέσουν κάτι για αυτά όλα. Κύριο Ντέιβις παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε και τον εισηγητή. Μία ερώτηση που θέλω να θέσω προς την Κομισιόν. Αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή όλο και περισσότερο έχουμε λιγότερου πόρου, του χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερο κλπ. Είναι θέμα το οποίο πραγματικά η Κομισιά τα έχει παρουσιάσει και έχει παρουσιάσει και αυτόν οδικό χάρτη. Και όταν φτάνουμε στην Αλία, μπορούμε να έχουμε περισσότερα ψάρια στι θάλασσέ μα και να αντιμετωπίσουμε τη ζήτηση σε αυτή την περίοδο της που είμαστε. Αλλά είναι σαφέ ακόμη του MSRY τη μέση ε, απόδοση, τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πραγματικά ποια είναι η κατάσταση, πώς είναι η δυνατότητα πραγματικά να υπάρξει νέα δυνατότητα από θεμάτων στις θάλασσές μας και τα πόσο αυτό θα είναι το καλύτερο τρόπος ή η καλύτερη οικονομική προσέγγιση του θέματος. Νομίζω πως η Κομισιόν μπορεί να διευκρινίσει ποια είναι η θέση της, ποιος είναι ο σκοπός της για την αναθεώρηση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Σκοπός είναι μόνο να σταματήσει την υπεραλίευση για να παραμείνουν τα αποθέματα σε, σε άνετο επίπεδο ή θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει μια στήριξη την οποία μπορεί να υποστηρίξει το, το μεγαλύτερο ποσοστό βεβαίω για να τη, για, στη που θα πρέπει να υπάρχει για την ανανεώση. Σε ευχαριστώ. Ο εκπρόσωπο της Κομισιόν έχει το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω πως όταν συζητήσαμε αυτά τα σημεία υπήρξαν μεγαλύτερες προηγηθικές όσον αφορά τη μεταρρυθμίση που πρέπει να γίνουν. Εξηγήθηκαν αυτά τα πράγματα πολύ σαφώς και είχαμε πολλές ώρες του Δεν υπάρχει αμφιβολία αυτή τη στιγμή πως η Κομισιό θέλει να δει το επίπεδο της εκμετάλλευσης, της θνησιμότητας για μέχρι το 2020. Η Κομισιόν εξάλλου ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει ούτε επιθυμητό είναι και δυνατό να ξεκινάμε να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή από το 2015 και μετά για δύο λόγους αυτό το πράγμα. Υπάρχει πολύ λίγη πληροφόρηση και επιστημονική επίσης για το θέμα των αποθεμάτων. Γνωρίζουμε βεβαίω ποια είναι η εκμετάλλευση η οποία γίνεται, αλλά δεν γνωρίζουμε τα άλλα δύο που σα είπα προηγουμένω. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια πρακτική στρατηγική επιλογή που θα πρέπει να γίνει. Ένα άλλο σημείο το οποίο πρέπει να υποθεί είναι ότι θα σκοπό εμείς, σαν στόχο, θα θέλαμε να έχουμε μια κατάσταση όπου τα αποθέματα που θα αποδίδουν ε, το μέγιστο όσο μπορούν. Εάν το εφαρμόσετε λοιπόν αυτό, τα στο μέγιστο επίπεδο του τα λιεύματα τα οποία παίρνονται από τη θάλασσα το, τότε, τότε εάν ε, τα αποθέματα θα αυξηθούν βεβαίω λαμβανομένες υπόψη πάντοτε και τη θυμόσια που υπάρχει και έτσι θα μπορεί να είναι πιο βιώσιμο το πράγμα σε σε 5-10 χρόνια από τη γνώση που έχουμε και τώρα θα μπορεί να επανέλθει στο επίπεδο το οποίο είναι το επιθυμητό. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο η Κομισιόν λαμβάνει μια στρατηγική θέση, λαμβάνοντα υπόψη την θεσιμότητα των ψαριών, των νυχθείων. Το δεύτερο σημείο είναι ότι θέλουμε ένα εργαλείο, ένα μέσο. Εάν δεν χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο, για αυτό το εργαλείο θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι τα αποθέματα τα οποία θέλουμε να θέσουμε, σε τι ποσό θα γίνονται και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να έχουμε αυτό το εργαλείο και είναι μια πρακτική επιλογή αυτή που πρέπει να κάνουμε σε αυτό το θέμα. Ένα πρόσθετο ακόμη σχόλιο έχει, είναι το εξή. Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά η Κομισιόν πρότεινα να φτάσουμε στα επίπεδα της εκμετάλλευσης θα πρέπει να αφήσουν τα αποθέματα να είναι πάνω από αυτό το οποίο έχει προβληθεί και θα πρέπει να γίνεται σε επίπεδα πιο κάτω από αυτά τα οποία έχουν προβληθεί. Αυτό γιατί η Κομισιόν πιστεύει πως είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την ασφαλιστική δικλίδα σε περίπτωση που συμβεί το απρόοπτο με τα αποθέματα και με την εκμετάλλευσή τους. Έτσι η Κομισιόν οικοδομεί αυτή την ασφαλιστική δικλίδα, για να υπάρξει αυτή η μακρο, ο μακροπρόθεσμος στόχος που έχει τεθεί για να φτάσουμε στο το αποτέλεσμα. Σε πιο σύγχρονα όρο θα έλεγα ότι τα επίπεδα αυτά είναι τα ανώτατα επίπεδα για την καλύτερη εκμετάλλευση των αποθεμάτων. Κάθε βήμα που κάνετε λοιπόν πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Κυρία Τόφη, έχει το λόγο παρακαλώ. Je remercie euh, la Commission pour, euh, pour ces précisions. Je constate que... Ευχαριστώ πάρα πολύ την Κομισιόν και θα πρέπει να δούμε ότι θα πρέπει να περιμένουμε μερικές μερικά θέματα τα οποία φαίνονται ότι δεν είναι πολύ σαφή, τα οποία έθεσε ο κ. Ντέιβις προηγουμένως. Για τα υπόλοιπα πιστεύω ότι είναι αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν όσον αφορά τη νέα πολιτική αλλίας και ο τερματισμός που θα γίνει τη συζήτησή μα για να έχουμε μια πλήρη συζήτηση για θέματα τα οποία έχουν εξεταστεί στα πλαίσια τη νομοδότηση. Πιστεύω να φώτισα ορισμένους προβληματικούς χώρους που πλούτησαν αυτό, αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ για τη συνδρομή των συναδέλφων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Τρότμαν. Να σας ανακοινώσω το ημερολόγιο τροπολογίες μέχρι τις 6 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι, ψηφοφορία στην Επιτροπή 24 και 25 Ιανουαρίου και ψηφοφορία στην Επιτροπή ΕΜΒΗ τον Απρίλη. Απρίλη, λάθος δεν μπορεί. Στην Επιτροπή ΕΜΒΗ λοιπόν η ψηφοφορία θα γίνει τον Απρίλιο. Εντάξει. Εμείς βιαστήκαμε λοιπόν. Ωραία. Κλείσαμε το 14 και περνάμε στο σημείο 15. Ο κύριος Λεβίν, ε, κύριο Λεβίν δεν σας είχα δει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που επιτρέπετε να... Διότι εκπλογήκαμε με, Ε, ψηφίσαμε για την ε, συμφωνία που έγινε με τη Βενεζουέλα. Είπατε, το συζητήσαμε αυτό στους συντονιστές. Μπορεί να μας εξηγήσετε γιατί δεν ψηφίσαμε για αυτό το θέμα. Αυτό που είπα είναι το εξή. Συμφωνήσαμε στους συντονιστές να προσφύγουμε στο δικαστήριο ε, εναντίον του Συμβουλίου. Δεν είπα τίποτα άλλο. Δεν ψηφίσαμε διότι η νομική υπηρεσία μου είπε πως αν πρόκειται να προσφύγουμε για κατάρριξη της νομοθετικής πράξης δεν χρειάζεται να ψηφιστεί σήμερα αυτή η πράξη στην Επιτροπή. Εγώ ακολούθησα απλώς τη σύσταση της νομικής υπηρεσίας. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα να το ξαναρωτήσουμε, να ξαναρωτήσουμε την νομική υπηρεσία. Εμένα η νομική υπηρεσία μου είπε πως αν πρόκειται να εκκινήσουμε την διαδικασία προσφυγής, κάτι το αποφασίσαμε σήμερα το πρωί, δεν είναι απαραίτητο να ψηφιστεί το θέμα αυτό, η πράξη αυτή στην Επιτροπή. Εγώ ακολούθησα την γνωμοδότηση αυτή. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, πέστε μου το και θα δούμε. Ζητήσαμε την γνώμη της, νομοθετικής, της ε, νομικής επιτροπής, ε, ε, της ε, νομική υπηρεσία. Και μας είπε αυτό που ακριβώς σα ανέφερα μόλι τώρα. Σημείο 15 τη διάταξη. Στρατηγική τη Ευρωπαϊκής Ένωση για την βιοπικιλότητα με ορίζοντα το 2020. Εισηγητής ο κύριος Ριβελίνη. Η Επιτροπή ΕΜΒΗ θα ψηφίσει την έκθεση αυτή στις 26 Φεβρουαρίου. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο λοιπόν. Γι' αυτό το λόγο ο εισηγητής θα μας υποβάλει κατευθείαν το προσχέδιο γνωμοδότησης. Κύριε Ριβελίνη, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Υπό την ιδιότητα του εισηγητού, καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος, τη Δημόσια Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, η οποία είναι αρμόδια για το λόγο θέμα, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματος που θα εγκρίνει ορισμένες υποδείξεις, ορισμένες προτάσεις, τις οποίες με την άδειά σας θα ήθελα εν συντομία να σας περιγράψω. Πρώτη πρόταση υπόδειξη. Υπογραμμίζω ότι κανένα κράτο μέλο δεν είναι θέση να διαχειριστεί το πρόβλημα τη απώλεια βιοπικιλότητος. Ειδικότερα στα θαλάσσια οικοσυστήματα και ότι οι κυβερνήσει των κρατών μελών οφείλουν να συνεργαστούν και να συντονίσουν τι προσπάθειε του κατά τρόπον πιο αποτελεσματικό προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ένα ζήτημα το οποίο είναι παγκοσμίου εμβέλεια και φύσεω. Δεύτερη υπόδειξη η πρόταση. Επισημαίνω ότι η ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής για την βιώσιμη ανάπτυξη του Ιωάννησμπουργκ του 2002, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεω προσυπέγραψαν τον στόχο επίτευξη μιας μέγιστη αηφόρου αποδόσεως, βιώσιμης αποδόσεως, για τα αποθέματα τα οποία θα έχουν μειωθεί μέχρι το 2015. Ωστόσο, καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει και να επανεξετάσει την προσέγγιση η οποία βασίζεται στην μέγιστη βιώσιμη απόδοση, λαμβάνοντας υπόψη της όλες τις πτυχές που χαρακτηρίζουν τον νυχτικό πληθυσμό και ειδικότερα τις διαστάσεις, τη διαστάση, την ηλικία, την κατάσταση αναπαραγωγής και αντιμετωπίζοντας έτσι και οριστικά το ζήτημα, θέλετε, των συνθέτων ε, αποθεμάτων από διαφορετικά είδη. Τρίτη υπόδειξη πρόταση. Υπογραμμίζω την σημασία το να διαθέτουμε επιστημονικές συμβουλές οι οποίες θα βασίζονται σε αξιόπιστα στοιχεία και πλήρη στοιχεία προκειμένου να μπορέσουμε να διακριθούμε αποτελεσματικά και με τρόπο βιώσιμο την αλεία. Κατά τα άλλα, προτείνω στο σημείο 4 προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω να αργοποιήσουν και να χρηματοδοτήσουν πλήρω τη νέα στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για την βιοπικιλότητα μέχρι το 2020, εξασφαλίζοντα ότι οτιδήποτε μέτρο χρηματοδότηση που θα ιδιωτηθεί θα συνάδει με τους σχετικούς νόμους για την προστασία της βιοπικιλότητος και των υδάτων. Ένα άλλο σημείο το οποίο θα ήθελα να σας προτείνω και να θέσω υπόψη σας ότι η επίτευξη των έξι στόχων της νέας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε ό,τι αφορά την βιοπικιλότητα μέχρι το 2020 εξαρτώνται από την τήρηση υφισταμένων διατάξεων που έχει ήδη δηλαδή θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον σωστό, αν θέλετε, συντονισμό των σχετικών προγραμμάτων. Ειδικότερα το δίκτυο των προστατευμένων ζωνών Natura 2000 και του προγράμματος Life Sin. Ο έκτο, η έκτη πρόταση της υπόδειξης, την οποία θα ήθελα να θέσω υπόψη σας, είναι ότι η πραγματική απόδειξη είναι και η δέσμευση την οποία ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση να πετύχει τους στόχους σε ό,τι αφορά την βιοπικιλότητα δεν πρέπει να εξατομικεύονται στα λιδινά στρατηγική, αλλά στις μελλονικές μεταρρυθμίσεις των κοινών πολιτικών γεωργίας και αλίας, όπως και στο πολιετές πλαίσιο το χρηματοοικονομικό. Υπενθυμίζω και επισημαίνω επίση ότι η επιτυχία της πρώτης στρατηγική οφείλεται στο γεγονός ότι η προστασία της βιοποικιλότητος δεν ήταν ε, αρκούντος ενσωματωμένη στις λοιπές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Καλό και αυτό είναι ένα άλλο σημείο τώρα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει δείκτες αξιόπιστους της βιωσιμότητας περιβαλλοντικής, περιβαλλοντικής αηφορίας και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την θαλάσσια βιωσιμότητα και την παράκτεια, προκειμένου να αξιολογήσει το επίπεδο της πρόοδου που θα έχει σημειωθεί προς την επίτευξη του πλήρους και συμπληρωματικού στόχου που είναι η προστασία της βιοποικιλότητας. Τέλος, Είμαι ικανοποιημένο και με ευχαριστεί ότι το, σχέδιο που παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο του 2011 αναπτύσσεται από τέσσερι οργανισμού τη Ευρωπαϊκή της Μεταξύ των οποίων ο ΦΑΟ, προκειμένου να, να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τη δέσμευση για να περιορίσουν τι απώλειε και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τι απώλειε που είναι η υπερβολική αξιοποίηση των πόρων, την ρήπανση και την απώλεια της βιοποικιλότητας. Πρόεδρε, και ευχαριστώ κύριε Ριβελίνη για την έκθεσή σας. Νομίζω ότι έχει πολλά καλά θετικά σημεία με τα οποία συμφωνούμε. Πιστεύω πάντως πως το σημείο υπαριθμών 8 που λέει προκειμένου να επιτευχθούν οι δεσμεύσει τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για δίποτε σε ό,τι αφορά του στόχου βιοπικιλότητα, πρέπει να ενσωματώσουμε του στόχου αυτού τόσο στην κοινή αγροτική πολιτική όσο επίση και στην κοινή πολιτική αλλία. Αυτό είναι κάτι που αποτελεί, αν θέλετε, το σημείο κλειδί στην όλη αυτή υπόθεση. Και βεβαίω είναι κάτι το, στο οποίο θα πρέπει να δίδετε έμφαση στην έκθεσή σας. Και χαίρομαι πολύ που το κάνετε αυτό και το πετυχαίνετε αυτό. Έχω βεβαίως κάποιες ερωτήσεις, τις οποίες θα ήθελα να σας θέσω. Ζητάτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει και να εξετάσει την προσέγγιση MSY, Αντιμετωπίζετε το ζήτημα, θέλετε, των αποθεμάτων πολλαπλών ειδών. Συμφωνώ μαζί σας ως προς χρειάζεται μια οικοσυστημική προσέγγιση. Και το συζητήσαμε αυτό μάλιστα σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου που έγινε για τα οικοσυστήματα και για τα regime shifts, για τις μετατοπίσεις δηλαδή, που, που θα πρέπει να ελέγξουμε συνολικά και να λάβουμε υπόψη μας το συνολικό στο οικοσύστημα. Διερωτώ με αν αυτό εννοείται μετά από θέματα πολλαπλών ειδών σε σχέση με το MSY ή αν έχετε κάτι άλλο κατά νου. Είναι δύσκολο πάντως να βγάλει κανείς νόημα από αυτά που γράφετε και αυτό που λέτε στην γνωμοδότησή σας. Ζητήσατε αξιόπιστα και πλήρη στοιχεία για αποτελεσματική και βιώσιμη διαχείριση της αλίας με τα πλήρη δεδομένα. Βεβαίως θα ήθελα και εγώ να τα έχω αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι η έλλειψη δεδομένων θα πρέπει να μας παρεμποδίσει από το να λάβουμε δηλαδή τις ορθές ε, αποφάσεις διαχείρισης και εφαρμόσουμε και την αρχή της προφύλαξης. Επομένως νομίζω ότι αυτή η αρχή της προφύλαξης είναι κατάλληλη και καλό θα είναι να αναφέρεται στο πλαίσιο αυτό. Έχω επίσης και ένα άλλο ερώτημα. Δεν το έχω ακόμη αυτό ελέγξει, αλλά αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα μέχρι το 2020, και ειδικότερα το στόχο 4 που αφορά στην βέλτιστη διαχείριση των ηχθικών αποθεμάτων. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό ο στόχος βαθμού 4. Και μιας και επίσης αναφέρεται συγγνωμοδότησή γνωμοδότησή σας τι δεσμεύσεις που είχε αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στην UNESCO, στον ΦΑΟ και στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, στον IMO δηλαδή, υπάρχει μια νέα περιβαλλοντική διάσκεψη που θα γίνει στο Ρίο Ντετζανέρο του χρόνου, Ρίο ΣΥΝ. Και νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια για να επηρεάσουν δηλαδή την ε, ημερήσια διάταξη και θα μπορούσαμε να βάλουμε την αηφορία των ωκεανών και τη βιωσιμότητα πάνω πάνω στην ημερήσια διάταξη ε, θα ήταν επιθυμητό. Γι' αυτό λοιπόν ίσως να χρειαστεί να καταθέσουμε κάποιες υπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Εκ μέρου τη Κομισιόν παρόν ο κ. Μπάξουτ από την ε, Γενική Διεύθυνση ΕΜΒΗ. Δεν είναι εδώ. Τον καλέσαμε, αλλά είναι απόν. Υπάρχει κανείς άλλος από τη Γενική Διεύθυνση ΕΜΒΗ που μπορεί να μας διαφωτίσει. Είμαι συντονίστρια και δεν μπορώ να λάβω θέση. Αλλά σε ό,τι αφορά τα θέματα αλληλεία, έχουμε ένα συνάδελφο από τη Γενική Διευθυνσία Αλληλεία, ο οποίο θα μπορούσε να σα πει λίγα λόγια. Eh, eh, Λυπάμαι που δεν έχουμε επαρκή εκπροσώπηση της Κομισιόν. Θέλετε να πάρετε το λόγο, θέλετε να πείτε κάτι. Α, το, το, το μπουκάλι είχατε στο χέρι σας. Οκ, okay, νόμιζα ότι ήταν το μικρόφωνο. Νο, νο, νο, νόμιζα ότι θέλατε να, να πάρετε το λόγο. Ε, λυπάμαι και διαμαρτύρομαι που η Κομισιόν δεν εκπροσωπείται επαρκώς. Ε, και δεν μας, έχουν, δεν μας έχει ενημερώσει η Κομισιόν και για ποιο λόγο ε, δεν ήρθε ο εκπρόσωπος που είχαμε καλέσει. Κύριε Ριβελίνη, έχετε το λόγο. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να προσθέσω θα ήθελα στα επιχειρήματα τα οποία ανέπτυξε η συνάδελφο Λουβίν προηγουμένω, ότι πιστεύω ότι ευθυγραμμίζονται, συνάδουν πλήρως δηλαδή με αυτά τα οποία ε, μίλησα προηγουμένω κατά 99%. Συμφωνούμε δηλαδή απολύτω. Απλώ να διευκρινίσω ένα σημείο θα ήθελα το οποίο έθεσε η συνάδελφος ή θέλησε να δώσει έμφαση η συνάδελφος στο σημείο αυτό. Θέλησα να υπογραμμίσω τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιοπικιλότητα μέχρι το 2020. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το στόχο 4. Γιατί μιλούμε για την αλληλεία αυτή τη στιγμή και πρόκειται για μέτρα τα οποία αφορούν και άπτονται τη αλληλεία. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να ασχοληθώ με την καλύτερη, την βέλτιστη διαχείριση αυτή των νυχτικών αποθεμάτων. Αυτό μου φαίνεται κάτι το αντικειμενικό επίσης, διότι είμαστε στην Επιτροπή Αλίας. Άρα, αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο θέλησα να υπογραμμίσω, να επισημάνω το σημείο αυτό. Κατά τα άλλα, συμφωνώ 100% μαζί σας. Κατά τα άλλα. Και παρόλο που δεν συνεννοηθήκαμε, την έκθεση αυτή τη συντάξαμε αυτήν δύο διαφορετικά άτομα. Δεν έχω τίποτα πάντως άλλο να προσθέσω. Ωραία. Τι μας μένει το χρονοδιάγραμμα, υποβολή τροπολογιών, ε, βιαζόμαστε γιατί θα ψηφιστεί στο τέλος Φεβρουαρίου στην ΕΜΠΗ. Συνεπώς 6 Ιανουαρίου, 12 ώρα το μεσημέρι, η προθεσμία για τις τροπολογίες. Η Επιτροπή μας θα ψηφίσει 24 και 25 Ιανουαρίου. Ωραία, κλείνουμε και το 15. Περνάμε στο σημείο 16. Απαλλαγή 2010, Γενικό προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τμήμα 3. Επιτροπή. Εισηγητή ο κύριο Μιλάνα. Θέλετε να πάρετε το λόγο εσεί ή να το δώσετε στην Κομισιόν πρώτα. Κύριε Μιλάνα, έχετε το λόγο. Πρόκειται για γνωμοδοτήσεω. ότι η γνωμοδότηση τη επιτροπή Κον. Δηλαδή πρόκειται για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Παρόλο που, παρόλο που είχαμε ήδη την ευκαιρία με την γραμματεία να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Η απαλλαγή του προπολογισμού γίνεται από το Κοινοβούλιο προκειμένου να αξιολογηθούν οι δαπάνες και αν δαπανήθηκαν όπως θα έπρεπε. Και βασίστηκα σε δύο στοιχεία. Την ποσότητα των δαπανών, το ύψος δηλαδή των δαπανών, και την αποτελεσματικότητά τους στην χρηματοδότηση και στην υλοποίηση των δράσεων. Και μετά από αυτή την ανάλυση θα μπορούσα να πω ότι συνολικά υπάρχει ένα στοιχείο αρκετά ικανοποιητικό, αρκετά ικανοποιητικό με τα αποτελέσματα προπολογισμού, δηλαδή για τη Γενική Διεύθυνση για τι θάλασσε, για τη Διεύθυνση ΜΑΡΕ, πέραν κάποιων ζητημάτων στα οποία θα αναφερθώ αργότερα. Γενικά το συλλογικό ποσοστό χρηματοδότηση εκτέλεση του προπολογισμού ήταν άνω των 97%. Πράγμα το οποίο να αυτό αποτελεί ένα καλό αποτέλεσμα. Φτάσαμε δηλαδή το 80% του 2010 των ποσών που είχαν διατεθεί. Και αυτό είναι καλό αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, για το συγκεκριμένο κεφάλαιο, το 1102 δηλαδή, το σχετικό δηλαδή με την αγορά της αλίας, είχαμε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο δαπανών, πράγμα το οποίο οφείλεται βασικά σε μια κατάσταση για την οποία κατά τη διάρκεια του 2010 δόθηκε, δόθηκαν χρήματα στις έξογος απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ του να γίνουν δεκτές κάποιες δαπάνες σχετικά με τις περιφέρειες αυτές. Μάλιστα μια πρόσθεση, πρόσφατη επαλήθευση που έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε νομίζω θετικά αποτελέσματα. Οδήγησε ο κατά για το 2010-2011 ξεπεράστηκαν τα προβλήματα με την αναστολή των, προ... πληρωμών δηλαδή. Και οι πληρωμές αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια του 2011. Βέβαια στο ποσοστό εκτέλεσης υπερ κατά τη δηλαδή το 70%. Πράγμα το οποίο καθόρισε και θα πρέπει να το δούμε αυτό κάπως καλύτερα και πληρέστερα και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα γίνει. 18 εκατομμύρια του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης δόθηκαν για το σκοπό αυτό. Και βεβαίω αυτό δεν είναι θετικό, δεν είναι ένα στοιχείο θετικό αναφορικά με τη διαχείριση. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο γύρεται και γέρθη και χάρη στην βέλτιστη τοποθέτηση των συναδέλφων του Ελεκτικού Συνεδρίου που έτέσε στη διάθεση της Επιτροπής μας. Και θέσαμε και ένα ζήτημα αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στο Ελεκτικό Συνέδριο ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το 2001 σχετικά με μια επένδυση η οποία έγινε στη Γερμανία για τον Γάβρο, για την Ατζούγια δηλαδή, και το πρόγραμμα του θα έπρεπε να κλείσει το 2011 και να έχει ολοκληρωθεί. Και το γεγονός ότι δεν ολοκληρώθηκε υπάρχουν επιφυλάξεις του ελεκτικού συνεδρίου και ερευνά αυτή τη στιγμή το ελεκτικό συνεδρίο την απάντηση που δόθηκε στο ερώτημα αυτό σε έντοφα χρηματοδότηση από τη Γερμανία. Πρόκειται για μια επένδυση που χρησιμοποίησε τα κέρδη σαν Πρόκειται δηλαδή για την κατασκευή, αν θέλετε, μια δημόσια εγκατάσταση που στη συνέχεια το εμπιστεύτηκε, το ενοικίασε δηλαδή σε ιδιώτες και χρησιμοποίησε δηλαδή τα ευρωπαϊκά κονδύλια, τους ευρωπαϊκούς πόρους, στο υψηλότερο δυνατό βαθμό για μια δημόσια επιχείρηση, αλλά στην πραγματικότητα η χρήση αυτή είναι καθαρό ιδιωτική. Εξετάζεται ακόμη αυτό το θέμα, ηγέρθηκε το του αυτό και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουν και πάρα πολύ αν θέλετε στην επιβεβαίωση. Έχει ξεπεράσει τα 5-6 χρόνια η έρευνα στην υπόθεση αυτή. Πρέπει βεβαίω να υπογραμμίσουμε ότι πρόκειται για μια διαδικασία η οποία, αν θέλετε, θα πρέπει να κλείσει νωρίτερα και στι επίσημε επαφέ που είχαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια των προσφάτων εβδομάδων μας εγγυήθηκε ότι βρισκόμαστε ακόμη στην τελική ευθεία. Ελπίζουμε να μην βρούμε αυτή την επιφύλαξη και στον, στην απαλλαγή αυτή που θα γίνει για το 2011, το προβλογισμό του 2011. Και συρωματικά μάλιστα βλέπουμε θετικά την εκτέλεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Ζήτησα, ζήτησα και σε σχέση πάντα με τις λοιπές μας δραστηριότητες ζήτησε να γνωρίζω εν λεπτομερία σε σχέση με τις αλληλευτικές συμφωνίες την, τις ψήφους για την τομεακή, τα κονδύλια για την τομεακή υποστήριξη. Και βεβαίω αυτό θα το δούμε με του συναδέλφου, θα ζητήσουμε με του συναδέλφου τη μεταρρύθμιση. Το 62% των πόρων που προορίζονταν για τι διεθνεί συμφωνίε, που είναι αν θέλετε πόροι που συνδέονται με την εμπορική συμφωνία και το 28% πρόκειται για πόρου οι οποίοι προορίζονται κονδύλια που προορίζονται να στηρίξουν τομεακά και αυτό είναι ένα δεδομένο, ένα στοιχείο το οποίο είναι ευκαιρία της ευάθυνσης σε ό,τι αφορά την απαλλαγή για το του 2010 είναι χρήσιμο και καλό θα ήταν και μας επιτρέπει να επιχειρηματολογήσουμε και σε σχέση με την... Ε, το πού θα δοθούν και θα διαλυθούν αυτοί οι πόροι. Επιβεβαιώνω επίσης και μια γνώμη που θα βάλουμε και στην γνωμοδότηση, που είναι ότι υπάρχει ανεγκαιότητα, σε ό,τι αφορά τις αλληλευτικές συμφωνίες, να υπάρχει η δυνατότητα να συμπεριλάβουμε και συμπληρωματικά και να παρακολουθούμε, αν θέλετε, τη διάρκεια και όχι μόνο το τέλος Κλείνω με το χρονοδιάγραμμα. Νομίζω ότι θα μπορούσα να σα παρουσιάσω ένα γραφό εργασία για την συνεδρία στι 27 Ιανουαρίου του 2012 και 27 Φεβρουαρίου δηλαδή για την κατάσταση των τροπολογιών. Θα έχουμε ένα, μήνα δηλαδή για να τροποποιήσουμε την γνωμοτότηση, η οποία θα είναι μια πολύ σφιχτή γνωμοδότηση, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στη ψηφοφορία στην Επιτροπή Αλίας στις 28 29 Φεβρουαρίου. Η προθεσμία είναι ο Απρίλιος, η συνεδρία στην Επιτροπή θα γίνει το Μάρτιο και θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Μαΐου. Ευχαριστώ επίσης τα μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου που είναι σήμερα παρόντα η οποία απήντησαν, τα οποία απήντησαν, αν θέλετε, σε πολλά email που του στείλαμε κατά τη διάρκεια τη περίοδου αυτή. Αλλά ευχαριστήσω και τη γραμματεία. Αλλά δεν βλέπω εδώ με πρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φτάνει. Θα φτάσει δηλαδή όταν θα έχω τελειώσει να μιλάω εγώ. Πολύ θετικό αυτό. Δεν ξέρω τι συνέβη ή θα μπορούσε να συμβεί. Ευχαριστώ πάντως. Θα δώσω τον λόγο στους εκπροσώπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τους ευχαριστώ που είναι εδώ. Είναι ο κύριος Έντουαρτ Φένεση. Ελπίζω να το προφέρω σωστά. Και ο κύριος Κονσιέλ. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο θέλει να πάρει το λόγο. Και οι δύο ενδεχομένω Σας ακούμε. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας καλέσατε. Δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να έρθουμε ενώπιν της επιτροπές και θα, ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πρόσκλησή του. Λέγομαι Edward Fantasy. Είναι διευθυντής της, του πρώτου τμήματος του Ελεκτικού Συνεδρίου και από των φυσικών πόρων βέβαια. Σε αυτό περιλαμβάνονται τα θέματα της αλληλείας και ότι άπτεται και της θάλασσας. Βεβαίω, η αλληλεία είναι ένα μικρό μέρος όσον αφορά τους πόρους του προϋπολογισμού. Όσον αφορά την νομιμότητα και τη θεμικότητα του θέματος, Ε, είναι στο μέσο που οποίο έχουμε περάσει αρκετά δύο-τρία χρόνια και ξέρουμε τι γίνεται και από το 10 και μετά έχουμε νέα περιπτώσεις που έχουν εξεταστεί με ελάσσονα θέματα τα οποία, τα οποία δεν είχαν μεγάλη επίπτωση και μεγάλα αποτελέσματα. Όσον αφορά τώρα τη μικρή σημασία που δίδουμε σε αυτό το θέμα δεν είναι ότι είναι αυτό καθ' ελάχιστη σημασία αλλά υπάρχουν χώροι που έχουν ε, με μεγάλα ποσά τα οποία διακυβεύονται και όπου είναι η αγροτικό τομέα με του φυσικού πόρου εκεί. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο, για τι λεπτομέρειε, θα περάσω το λόγο στον κύριο Κορφίλ, ο οποίο θα σα θα σας δώσει μια μικρή περίληψη για τα θέματα τα οποία εξετάσαμε και αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια αυτή τη του ελέγχου των οποίων κάναμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ο μου είπε πρώτα θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και εγώ γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα να πούμε. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα για φέτος και μόνο για όσον αφορά την απόρριψη μιας επιφύλαξης η οποία είχε η, για τις για είναι με επιφύλαξη την οποία έχει η Κομισιόν από αρχές από το 2009 είναι το μόνο σημείο το οποίο έχουμε εισαγεί στην έκθεσή μας την ελεγκτική όπως ο διευθυντής μου είπε υπήρξαν 239 ε, δικαιοπραξίες οι οποίες έγιναν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έγιναν από πολίτες για να σας δώσω όμως μία ιδέα αυτού του πράγματα τίποτα πολύ σημαντικό για παράδειγμα οι τοπικές αρχές αρχές μερικές φορές ζήτησαν πάρα πολλά ε, βάρη η ποσά τα οποία έβαλαν ήταν ελάχιστη ε, σημασία σε όλα αυτά τα οποία εξετάστηκαν και δεν έχουν ιδιαίτερα βάρο, ωστόσο ελέγχθησαν. Όσον αφορά την ομιμότητα αυτών των ε, δικαιοπραξιών δεν υπάρχει τίποτα να υπογραμμιστεί εκτός από μερικά ελάσσονα τα οποία βεβαίως έχουμε υποβάλει προς, προς αρμόδιες αρχές της Κομισιόν. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που ήρθατε μέχρι εδώ και για τις παρατηρήσεις σας. Ο κύριος Γιόνσον, Τζόνστον μόλις έφτασε, δεν με ακούει, αλλά μόλις έφτασε. Κύριε Τζόνστον, λέω ότι μόλις φτάσατε, σας καλωσορίζω. Ε, μόλις που προλάβατε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Ε, περιμένουμε θα συζητηθεί αργότερα το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά τι διαδικασίε απαλλαγή. Νομίζω ότι στο κεφάλαιο 3 της αιτήσιας έκθεσης του ε, Ελεκτικού Συνεδρίου ε, γίνεται σαφές ότι σε ό,τι αφορά το θέμα της αλλίας και των θαλασσιών υποθέσεων δεν υπάρχουν σημαντικά ζητήματα και προβλήματα. Αυτό βέβαια ε, δεν ελαχιστοποιεί τα ζητήματα τα οποία εντόπισε το Ελληνικό συνέδριο. Ε, ήδη μας ε, έδωσε ο εκπρόσωπος του Ελληνικού συνεδρίου ένα παράδειγμα. Για το θέμα της επιλεξιμότητας, ιδιαίτερω η Κομισιόν θα ε, λάβει τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που εντοπίστηκαν και θα φροντίσουμε έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητε διορθώσει από το εμπλεκόμενο κράτο μέλο. Σε ό,τι αφορά τι επιφυλάξει ε, εκ μέρου τη Κομισιόν, στι οποίε αναφέρθηκε το Ελληνικό Συνέδριο, να σα πω ότι παρακολουθούμε πάρα πολύ καλά τι επιφυλάξει. Θα αναλάβουμε την κατάλληλη δράση και θα ενημερώσουμε πλήρω για τις δράσεις μας στην δική μας ετήσια έκθεση του 2011. Τέλος, να πω δύο λόγια για την εκτέλεση του προπολογισμού. Ε, παρακολουθώ τα, ε, μάλλον διάβασα τα νούμερα για φέτος και με χαρά μου μπορώ να σας πω ότι το ποσοστό εκτέλεσης σε ό,τι αφορά δεσμεύσεις και πληρωμές είναι υψηλότερο το 2011 από αυτό το 2010. Όλα αυτά τα παρακολουθούμε πολύ στενά, ιδιαίτερα δεδομένων των δύσκολων οικονομικών συνδικών τις οποίες βιώνουμε. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι ε, οι εκταμιεύσεις γίνονται γρήγορα, διατηρώντας όμως τα επαρκή επίπεδα ελέγχου των δαπανών μας που επιβάλλονται. Ευχαριστώ. Κύριε Μιλάνα, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Δύο μικρό πράγματα. Τα είπατε σωστά. Νομίζω πως ό,τι είπατε αντιστοιχούν και η δική μας γνωμοδότηση θα είναι πάρα πολύ θετική. Παρόλο που θα επισημαίνονται τα ζητήματα τα οποία, όπως είπα στην αρχή, είναι κάπως προβληματικά. Αλλά σε σχέση με αυτά τα οποία είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να πω κι εγώ κάτι. Εμείς φέτος είχαμε προβλήματα σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Και δεν βρίσκουμε και δεν βρήκαμε του πόρου για να την χρηματοδοτήσουμε αυτή την ε, ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και η δική μας η πρόεδρος ε, έγραψε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δει πού βρίσκονται τα χρήματα, πού θα βρεθούν τα χρήματα για τη χρηματοδότηση ένα τομέα που το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι είναι στρατηγική σημασία για να μπορέσει να βοηθηθεί ο τομέα. Μιλούμε για λίγα εκατομμύρια ευρώ. Λίγα εκατομμύρια ευρώ. Για το 2011. Δεν αφορά το ζήτημα αυτό το δί, που δόθηκαν κάποια εκατομμύρια στα κράτη-μέλη. Εν πάση περιπτώσει δέχομαι αυτά τα οποία είπατε και χαίρομαι που το ποσοστό εκτέλεση του 2011 είναι πολύ ψηλό. Και θα ζητήσω να είμαι ε, και εισηγητή δηλαδή για την απαλλαγή του 2011 για να επαληθεύσω αν κατά τύχη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έδωσε τα χρήματα για την ε, ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Ζήτησε και μια έκπτωση 10 εκατομμυρίων ευρώ και επιστρέψαμε στα κράτη-μέλη τα χρήματα που του αναλογούσαν. Και αυτό θα ήταν, αν θέλετε, κάπω ε, άσχημο. Γι' αυτό λοιπόν θα ζητήσω από την πρόεδρο να είμαι και του χρόνου ε, αρμόδιος για την ε, απαλλαγή του 2011. Εξαιρετικά. Επόμενη συνεδρία, στην επόμενη συνεδρίαση θα δούμε το προσχέδιο γνωμοδότησης. Ευχαριστώ του κύριους ε, από το Ελεκτικό Συνέδριο, από την Κομισιόν, τον κύριο Τζόνστον και τον κύριο Μιλάνα. Περνάμε στο υπαριθμό 17 σημείο της Μέσιας διάταξης, απαλλαγή 2010, κοινοτική υπηρεσία ελέγχου της αλίας. Εισηγητής ο κύριος Χατζημαρκάκης, ο οποίος είναι απόν. Λυπάμαι που δεν είναι εδώ. Οπότε να βάλουμε τη συζήτηση. Κρίμα που δεν είναι εδώ οι, οι βουλευτές όταν πρέπει να είναι για να συζητήσουμε το θέμα τους. Περνάμε στο 18, διάφορα, υπάρχει καν μια ε, Κάποιο θέλει το λόγο, όχι. 19 ανακοινώσει τη Προέδρου σχετικά με τι αποφάσει που έλαβαν οι συντονιστέ. Νομίζω ότι σα μοιράσαμε ένα σημείωμα με τι αποφάσει που ελήφθησαν. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, απορίε κλπ. υιοθετούνται οι αποφάσει αυτέ. Σημείο 20. Προσεχή συνεδρίαση 24 και 25 Ιανουαρίου Ε, αυτά, καλές γιορτές, ε, ευτυχισμένος ο καινούριο χρόνος ε, και ελπίζω να τα ξαναπούμε το Γενάρη όλοι εδώ. Γεια σας.